Καλωσορίζω. Άρχεται η συνεδρίαση. Καλωσορίζω επίσης στο Κοινοβούλιο τον Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας πρώην προεδρεύοντα του Συμβουλίου και της προηγούμενης Προεδρίας καθώς και τον πρόεδρο Χωρός Μανουέλ Μπαρόσο και τον αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς της Επιτροπής. Πρώτον, θέμα στην ημερήσια διάταξή μας η Ουγγρική Προεδρία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρωθυπουργό Βίκτορα Ορμπάν, εξ του Συμβουλίου. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.